προσκαλούσα όσους συμμετάσχουν στην ώρα ερωτήσεων να έρθουν και να καθίσουν στα έδρανα στις πρώτες σειρές ε, στην Ολομέλεια. Η πρώτη ερώτηση στην ημερήσια διάταξή μας ε, σήμερα είναι ουσιαστικά μια κοινή συζήτηση, μια κοινή απάντηση από πλευράς Υπουργού. Ελπίζω σε τρεις ερωτήσεις από τον κύριο ρέχα, από τον κύριο Πόσετ, Χόρατσεκ, Πόσετ και Κελάμ. Και οι τρεις αυτές ερωτήσεις αφορούν την δικαιοσύνη, το σύστημα απονομής δικαιοσύνης και το κράτος δικαίου στη Ρωσία. Μπορώ να πω κύριε Υπουργέ ότι τώρα θα έχετε τον λόγο για να απαντήσετε ε, την πρώτη ερώτηση. Παρακαλώ. Ναι. Σας ευχαριστώ. Γνωρίζω ότι ο φίλος μου Μίλαν Χόρατσεκ που έχει διατυπώσει την πρώτη ερώτηση είναι ένα άτομο που επί μεγάλο χρονικό διάστημα καταβάλει προσπάθεια να παρακολουθήσει την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Ρωσία και θέλω να τον ευχαριστήσω για αυτό το περιεχόμενο αυτής της ερώτησης που αφορά ακριβώς αυτό που αυτό το σώμα θα έπρεπε να παρακολουθεί και να κάνει. Σε σχέση με την ερώτηση συγκεκριμένα τώρα, όσον αφορά το συγκεκριμένο εξειδικευμένο αυτό το θέμα θα ήθελα να τον διασφαλίσω ότι πλήρως συμμερίζεται το Συμβούλιο της ανησυχίες του για τις εξελίξεις όσον αφορά το κράτος δικαίου και την δημοκρατία στη Ρωσία. Το Συμβούλιο θεωρεί ότι η εταιρική μας σχέση με τη Ρωσία θα πρέπει να βασίζεται στον σεβασμό για το διεθνές δίκαιο τις αρχές ε, του κράτους δικαίου, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και γι' αυτό το Συμβούλιο θα συνεχίσει να ασκεί πιέσει επί της Ρωσίας να υλοποιηθούν πλήρως οι υποχρεώσεις που έχει υπογράψει και έχει επομιστεί η Ρωσία ως μέλος του Συμβουλίου της Ευρώπης και φυσικά ως μέλος ε, του ΟΑΣΕ. Και μέσα στο πλαίσιο επίσης της ε, PCA, της ε, Συμφωνίας ε, Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας με την ΕΕ. Η συγκεκριμένη περίπτωση που αφορά το ερώτημά σας και των συναδέλφων σας μας ανησυχεί ιδιαίτερα. Το Συμβούλιο θα συνεχίσει λοιπόν να παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς τα τεκτενόμενα στη Ρωσία τις ανησυχίες αυτές που έχει το Συμβούλιο όσον αφορά τη Ρωσία τις επαναλαμβάνει σταθερά μέσα στο πλαίσιο του πολιτικού διαλόγου και ιδιαίτερα μέσα στο πλαίσιο των διαβουλεύσεων για τα ανθρώπινα δικαιώματα που ξεκίνησαν το Μάρτιο 2005 ως πρωτοβουλία. Η Ρωσία σχετικά και σε σχέση και με άλλους τομείς οι θέσεις τους θα ληφθούν υπόψη σε σχέση με μια νέα συμφωνία με τη Ρωσία. Πολύ σημαντικό αυτό και επίσης ε, και υπό άλλες τυχές ε, των σχέσεών μας με τη Ρωσία το να επιτευχθούν ε, οι διατάξεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα σε σχέση με τη Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας Υποδιαπραγμάτευση είναι μία από τις προτεραιότητές μας όπως ε, αφορά άμεσα και τις διαπραγματεύσεις αυτές ε, όπως εγκρίθηκαν από την εντολή σε σχέση με το Συμβούλιο πέρυσι. Η στρατηγική σχέση εταιρική σχέση με την Ρωσία για την οποία κάνουν λόγο κάποιοι θα πρέπει να θεμελιώνεται στις αμοιβέ κοινά αναγνωρισμένε αξίες. Διαφορετικά δεν θα είχε νόημα. Χρειάζεται αυτή τη νέα συμφωνία η ΕΕ. Εξίσου τη χρειάζεται όμως και η Ρωσία. Είναι κέρια σημασία οι διαπραγματεύσει, όπως επίσης και το κείμενο της ίδιας της συμφωνίας για τις τα ανθρώπινα δικαιώματα και το κράτος δικαίου να είναι σεβαστές αρχές. Εγώ προσωπικά θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι η ενιαία στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι απόλυτα αναγκαία για να επιτύχουμε αποτελέσματα όσον αφορά τους Ρώσους. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Υπουργέ. Με την κοινή ερώτηση θα ήθελα να δώσω την ευκαιρία σε κάθε ένα από αυτούς που διατύπωσαν ερωτήσεις να διατυπώσουν μια επερώτηση σε ένα πρόσθετο διάστημα μισού λεπτού, ο ένας μετά τον άλλο. Και μετά θα ζητήσω από τον Υπουργό να απαντήσει σε μια πλήρη τοποθέτηση επί των τριών παρεμβάσεων. Έχει τον λόγο λοιπόν τώρα ο κύριος Χόρατσεκ πρώτο. Σας ευχαριστώ. Λειτουργεί αυτό. Ναι, λειτουργεί. Έχω ένα συγκεκριμένο κάποιο πρόβλημα, διότι στο παρελθόν επανειλημμένα από το Συμβούλιο μας δινόταν η απάντηση ότι λέει η προτεραιότητα είναι φυσικά οι σχέσεις μας με τη Ρωσία κτλ. κτλ. Όμως ακριβώς Στη συγκεκριμένη αυτή η περίπτωση όσον αφορά το πρόβλημα Χοντορκόφσκι για παράδειγμα του Λιέμπεντεφ και της ε, κυρίας Μάχτινα δεν έχει σημειωθεί καμία πρόοδος. Now, Τώρα ο κύριος παρακαλώ. Σα εκτιμώ ιδιαίτερα. Είσαστε ένα πεπειραμένο υπέρμαχος των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Εκτιμώ ιδίω ε, και την, ε, τον εφάνταστο χαρακτήρα και τη δημιουργικότητα των Τσέχων. Γι' αυτό ερώτησή μου, μπορείτε να μας βοηθήσετε να βρούμε νέου διάβλου ώστε μετά από πολλά χρόνια διακηρύξεων να οδηγηθούμε πιο κοντά σε μια επίλυση του προβλήματος, να υπάρξει κάποιος ακτιβισμός και τα θέματα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων χειροπιαστά έμπρακτα στις διαπραγματεύσεις με τη Ρωσία να βρεθούν αυτά περισσότερο στο επίκεντρο από ό,τι ήταν μέχρι τώρα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πόσελτ, ο κύριος Κέλαμ. Σας ευχαριστώ Υπουργέ για τις απαντήσεις σας. Αλλά συμφωνείτε ότι αν το Συμβούλιο είχε έντονα και πιστικά παρουσιάσει αυτό το πρόγραμμα προ τη ρωσική πλευρά, αποδεικνύοντας πως η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι σοβαρή σε σχέση με τέτοιες σκανδαλώδει παραβιάσει της δικαιοσύνης και οι οικονομικές σχέσεις θα βρίσκονταν σήμερα σε σωστότερη βάση. Συμφωνείτε ότι το τουλάχιστον ότι αν η αν δεν βρεθεί σωστή λύση στις υποθέσεις Χοντορκόφσκι και Μπάσμινα, ε, θα, ε, δεν πρόκειται η Ρωσία να σεβαστεί τις δεσμεύσεις της. Κοιτάξτε. Δεν μπορείτε να περιμένετε η τσεχική προεδρία να μείνει σιωπηλή και δεν σιώπησα για την κρίση, δεν ε, σιώπησα ούτε και για τις υποθέσεις Φοντορκόφσκι και άλλες υποθέσεις. Ε, θα ξέρετε ίσως ότι έχουμε συνεδρίαση τη Στρόικα το Φεβρουάριο και η Προεδρία θα την προσωπευθεί από τον Υπουργό Εξωτερικών Κάρος Σβάρτσεμπερκ και στις περιπτώσεις όπου ζητάμε, όπως για παράδειγμα για την κυρία Μπακούμινα, θα, σκεφτούμε τι βήματα θα ακολουθήσουμε, αλλά φυσικά είτε υπάρχουν αποτελέσματα ή όχι. Αυτό εξαρτάται από τους Ρώσους. Εμείς μπορούμε απλώς να φτιάξουμε κάποιο περιβάλλον, συγκεκριμένη ατμόσφαιρα, να πιέσουμε, αλλά από τους Ρώσους εξαρτάται αυτά τα αποκριθούν. Ερώτηση από τον κύριο Χάναν. Ευχαριστώ κύριε. Θα ήθελα να καλωσορίσω τον Υπουργό και να συγχαρώ την Τσεχική Προεδρία για την έναρξή της αλλά σοκαρίστηκα επίσης από ορισμένε ερωτήσεις συναδέλφων προς τον Τσέχο Προεδρεύοντα όπως ο κύριος Ντερόσα που είπε να αποσύρει την δήλωσή του ότι ίσως η συνθήκη της Λισαβόνας να μην είναι ακριβώς αυτό που αναμένουμε. Ναι, αλλά ποιο είναι το ερώτημα, λέει η Πρόεδρος εδώ μέσα. Παρακαλώ, τελειώσατε και δεν θέσατε ερώτημα. Συνεχίζει ο βουλευτής με κομμένο το μικρόφωνο. Και τώρα, επόμενο ερώτημα στην ημερήσια διάταξη. Ήταν της κυρίας Χάρκιν αλλά έχει αναλυφθεί από την κυρία Μακίνες. Ορίστε κύριε Υπουργέ μου. Κοιτάξτε. Σας ευχαριστώ μεν πολύ για αυτή την συγκεκριμένη ερώτηση γιατί προέρχομαι από μια χώρα που είναι μεγάλος υπέρμαχος του ελευθέρου εμπορίου 80% του ΑΕΠ μας προέρχεται από εμπορικές δραστηριότητες. Μπορείτε λοιπόν να είστε βέβαιοι ότι η Προεδρία μας θα παραμείνει προσιλωμένη στο στόχο της εξισορρόπησης, της εξέβρεσης μάλλον μιας ισορροπημένης συμφωνίας στον γύρο Ντόχας Πόε. Όσο για το θέμα των φιλοδοξιών της Προεδρίας μου, λέει ο μιλητής, έχουμε πει ποιες είναι οι προτεραιότητές μου. καθώς και τις προτεραιότητες του 18 μήνου προγράμματος του Συμβουλίου, όχι μόνο για την Τσεχική αλλά και για τις επόμενες προεδρίες. Σύμφωνα με το πρόγραμμα αυτό, η εμπορική πολιτική παραμένει πολύ σημαντικό εργαλείο για να λυθούν να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις της παγκοσμιοποίησης και για να προωθηθεί η οικονομική ανάπτυξη, θέση εργασίας και η ευημερία για όλους και όλες στην Ευρώπη. Θέλουμε να προωθήσουμε μια ανοιχτή οικονομία της αγοράς προς όφελος όλων. Η εμπορική πολιτική επίσης θα συμβάλλει στην επίτευξη των κλιματολογικών και περιβαλλοντολογικών στόχων της Ένωσης. Η Ένωση παραμένει προσιλωμένη στην επίτευξη μιας σφαιρικής συμφωνίας στον ΠΟΕΝΤΟΧΑ. Three priorities areas for its presidency of the Council Έχουμε και τρεις ακόμη στόχους. Μία από αυτούς, ένας από αυτούς είναι My country will highlight the importance of trade. Ε, ακριβώς η χρησιμοποίηση της εμπορικής ε, πολιτικής για την επίτευξη μεγαλύτερης ευημερίας και περισσότερων θέσεων απασχόλησης στα πλαίσια του στόχου που λέγεται Σφαιρική Ευρώπη. Η τσεχική δημοκρατία θα θελήσει να συνάψει και συμφωνίες με επίλεκτους εταίρους όπως το Μερκοσούρ, η Κορέα και η Ινδία, χώρες της Λατινικής Αμερικής, και την Κίνα, και να θα διαπραγματευτεί και εμπορικές συμφωνίες με τους ε, κοντινότερους ε, γείτονές μας όπως στην Ουκρανία. Το πρόγραμμά μας για τα εμπορικά θα το παρουσιάσουμε στις 20 Ιανουαρίου. Για την ασφάλεια των τροφίμων η Προεδρία φρονεί ότι ο παραγωγισμός δεν είναι η μόνη λύση. Γι' αυτό υποστηρίζουμε την απελευθέρωση του παγκοσμίου εμπορίου μέσα στα πλαίσια του DDA και οι συζητήσεις για τι μεταρρυθμίσεις της ΚΑΠ πρέπει να καταλήξουν σε μια πιο ανταγωνιστική οικονομία. Περισσότερες εξαγωγές. Αυτά είναι η βάση για τη βελτίωση της κατάστασης και ως προς την ασφάλεια των τροφίμων, η οποία αφορά πολύ βέβαια και το διεθνές εμπόριο τροφίμων γιατί χορηγεί φτηνότερα τρόφιμα στην αγορά. Η ασφάλεια των τροφίμων σήμερα δεν σημαίνει μόνο τοπική παραγωγή των τροφίμων, αλλά και την κατάλληλη χρηματοδότηση των εισαγωγών, αγκαίων εισαγωγών μέσω της εξαγωγής άλλων αγαθών. Ίσως αυτή να είναι η καλύτερη εγγύηση για τη δημιουργία μιας σταθερής προσφοράς. Ευχαριστώ κύριε Μαγκίνες. Ευχαριστώ για την λεπτομερή αυτή απάντηση που θα χρειαστεί να την μελετήσω. Πάντως εδώ έχει εγκριθεί μια έκθεση για την ασφάλεια των τροφίμων όπου λέγαμε ρητά ότι η αγορά δεν αρκεί για να δημιουργήσει την ε, τροφιμική ασφάλεια. Μπορείτε λοιπόν να μου εξηγήσετε αν πιστεύετε ότι το ελεύθερο εμπόριο είναι ο μόνος δρόμος. Αυτή είναι η προτεραιότητά σας. Ευχαριστώ. Ναι, να σας τα πω απλά, ναι. Αν υπάρχει ελεύθερο εμπόριο στη Γεωργία δεν είναι πρόβλημα αυτό. Είναι καλό πράγμα. Δύο ακόμη πρόσθετες ερωτήσεις, Πόσελτ και Καμάου. Πρώτα όμως Πόσελτ. Κύριε Υπουργέ, πάντα αναφέρεται η πολιτική για τη Γεωργία είναι για 3%, 3% όμως γεωργών. Υπάρχουν 100% όμως που καταναλώνουν τα τρόφιμα και εγώ ένας από αυτούς. Πιστεύω ότι η ασφάλεια η επισητιστική είναι ζωτική σημασία. Βλέπουμε τα προβλήματα σε σχέση με την εξάρτηση με ενεργειακά προϊόντα. Είμαι υπέρ του ελεύθερου παγκόσμιου εμπορίου. Πρέπει όμω να μπορούμε να τροφοδοτούμε με προϊόντα επισητιστικά τι ανάγκε μα και δεν μπορούμε να αφήσουμε όλε τι δομέ στην αγορά. Ευχαριστώ. Ο κύριο Καμάλ, παρακαλώ. Uh, Σα ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Καταρχήν, όπως και ο συνάδελφος πριν από μένα, ο κ. Χάναν, θα ήθελα να καλωσορίσω την Τσεχική Προεδρία. Ενδιαφέρουσα αντίθεση με την τελευταία Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ήθελα να ζητήσω συγγνώμη για την τροπιαστική συμπεριφορά ορισμένων συναδέλφων εδώ στην αίθουσα, ε, στο ημικύκλιο. Θέλω να σας ρωτήσω. Με αυτές τις εκλογές που θα γίνουν, Πώς θα ξεκινήσουμε τις διαπραγματεύσεις του ΠΟΕ. I think on the CAP reform, among those who Υπάρχουν ε, άνθρωποι που προσπαθούν να οθήσουν την, την Κομισιόν αυτή τη νέα πρόταση για τη μεταρρύθμιση του προπολογισμού, το λευκό βιβλίο. Προσπάθησα μάλιστα να διοργανώσω μια είδους, κάποιο είδους ε, συνεργασία με τον συνάδελφο του τη γιατί το 2009 είναι η Σουηδική και η Τσεχική Προεδρία και έχουμε παρόμοιες απόψεις. Πρέπει να ζητήσουμε για την υποβολή νομοθετικής πρότασης και φίλε μου, Πόσελτ, ξέρεις βέβαια, ότι έχουμε παρόμοια κουλτούρα και υπόβαθρο, και εμείς οι δυο είμαστε τα ζωντανά παραδείγματα ότι δεν υπάρχει πείνα στην Ευρώπη. και ότι ε, ε, η ευρωπαϊκή αγορά είναι καλή. Κάποια πολύ νόστιμα προϊόντα επίσης θα πρέπει να τα διατηρήσουμε στην Ευρώπη, όπως η βαρεζική και η τσεχική μπύρα. Και να μείνουμε ε, να καταναλώνονται τόσο στην Ευρώπη όπως και στην υπόλοιπο κόσμο. Περνάμε στο επόμενη ερώτηση για το μέλλον της κοινή γεωργικής πολιτικής. Υπουργέ. Yeah. Oh, Εδώ ερώτημα για την ΚΑΠ. Το Συμβούλιο κυρίε και κύριοι θα ήθελε να υπενθυμίσει ότι μέσα στο πλαίσιο της πολιτικής συμφωνίας που επετέφθη για την ενδιάμεση αναθεώρηση της ΚΑΠ από το Συμβουλίου στις 20 Νοεμβρίου 2008 είχε συμφωνηθεί από κοινού μια δήλωση Συμβουλίου και Επιτροπής μέσα στο πλαίσιο της συζήτησης που είχε ξεκινήσει στο Ανεσί της Γαλλίας στις 23 Σεπτεμβρίου για το μέλλον της ΚΑΠ μετά το 2013 και χωρίς ε, να ε, επηρεαστούν οι νέες δημοσιονομικές προοπτικές για την περίοδο αυτή δεσμεύονται το Συμβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξετάσουν εκ του σύνεγγυ τι δυνατότητε για την ανάπτυξη και διαμόρφωση των άμεσων πληρωμών στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα και την αντιμετώπιση του επίπεδου, διαφορετικού επίπεδου πληρωμών μεταξύ διαφορετικών κρατών. Θα μπορούσα να σας πω ότι η, η ενεξελίξη τσεχική προεδρία αυτό που θα κάνει είναι έχει την πρόθεση να διοργανώσει τη συζήτηση αυτών των θεμάτων στο άτυπο πλαίσιο υπουργικής συνάντησης, δηλαδή Υπουργών Γεωργίας που θα διεξαχθεί στο Μπρνο της Τσεχίας τον Μάιο 2009 και ο συνάδελφος στην κυβέρνηση υπουργό Γκαντάλοβιτς προσβλέπει στην εξέλιξη αυτής της συζήτησης. Στόχος μας είναι να διεξαχθεί μια συζήτηση για το μέλλον της ΚΑΠ και να την συντονίσουμε εξετάζοντας ε, τις δυνατότητες των γεωργικών πολιτικών εργαλείων στο επίπεδο των άμεσων πληρωμών που θα επιτρέπει μια μη αρνητική μεταχείριση, μη κριτική μεταχείριση έναντι των κρατών μελών και την χρήση των κονδυλίων των φορολογουμένων σε σχέση με την ΚΑΠ με τον πιο δίκαιο τρόπο, ενισχύοντα φυσικά την ανταγωνιστικότητα των Ευρωπαίων Γεωργών και βελτιώνοντα τη θέση τη Ευρωπαϊκή Γεωργία και ε, βιομηχανία τροφίμων σε μια παγκοσμιοποιημένη οικονομία τη αγορά, βελτιώνοντα την ποιότητα των γεωργικών προϊόντων φυσικά και λαμβάνοντας υπόψη ε, και τα θέματα που δεν εμπλέκουν με την αγορά καθώς επίσης και την αηφόρο ανάπτυξη της υπαίθρου. Η έκβαση αυτού του διαλόγου θα έπρεπε να οδηγήσει στην προλίανση του των όρων και προϋποθέσεων για μια εξυγχρονισμένη ΚΑΠΑ με ίσους όρους και προϋποθέσεις και το υπογραμμίζω αυτό για όλα τα κράτη-μέλη. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ τον Προεδρεύοντα για την απάντησή του και θέλω να τον ρωτήσω σε σχέση με τα προγράμματά τους κατά τη διάρκεια της Τσεχικής Προεδρίας πώς προτίθεται να βοηθήσουν τις της περιοχές πώς προτίθεται να τις υποστηρίξουν γιατί εγώ κατάλαβα ότι αυτές οι περιοχές είναι που εμπίπτουν στην δικαιοδοσία της ΚΑΠ. Θα ήθελα, θα να ξέρω ακριβώ τι πρόκειται να κάνει σε αυτό το θέμα, Υπουργέ. Νομίζω, προσέξτε, το πρόβλημα των μειονεκτικών περιοχών στην Ευρώπη πανευρωπαϊκά είναι ένα ιδιαίτερο πρόβλημα που διαρκώς συζητείται στο πλαίσιο της ΚΑΠ και θα έλεγα ότι όλοι οι περισσότεροι συμφωνούμε ότι θα έπρεπε να κινηθούμε από το, επίπεδο, από το πλαίσιο άμεσων πληρωμών στις πληρωμές μέσω ενός πλαισίου ανακατανομής για την ανάπτυξη της υπαίθρου και του τοπίου αντί να συνεχίσουμε μέσα σε προστατευτικά μέτρα και παρεμβάσεις. Υπάρχουν λοιπόν εργαλεία και μέσα να επιτευχθεί αυτό και σίγουρα θα έλεγα συνεργαζόμαστε από, ε, εκ του σύνεγγυς με την Επίτροπο Fisher Boyle για να ευδοκιμήσει αυτός ο στόχος και σίγουρα θα υπάρχει η δυνατότητα να προσεγγιστεί επίσης ε, και ο ειδικός μας Υπουργός ε, Γεωργίας και να συζητηθούν αυτά τα θέματα πιο εξειδικευμένα με αυτόν. Έχω διάφορα αιτήματα για υπερωτήσεις θα πάρουμε εκείνους τους ευρωβουλευτές που δεν παρενέβησαν. Κυρία Ντόιλ, πρώτα η κυρία Ντόιλ παρακαλώ. Thank you. May I... Uh, Σας ευχαριστώ. Εύχομαι στην Ιδρυτική Προεδρία κάθε επιτυχία κατά τη διάρκεια της θητείας σας. Θα ήθελα ο υπουργό να σχολιάσει την εμπειρία των Τσέχων γεωργών ε, στην τσεχική βιομηχανία γεωργίας και τροφίμων να μας πούν ε, αν είναι ικανοποιημένοι μέχρι στιγμή και αν ήταν βελτίωση κάπου για εκείνους. Πώς βλέπετε εσείς λοιπόν την ε, κοινή γεωργική πολιτική. Να ακούσουμε και την ερώτηση της κυρία Τικάου. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Δυστυχώς η οικονομική κρίση οδηγεί σε απώλεια θέσεων απασχόλησης. Η αγοραστική δύναμη μειώνεται. Η ποιότητα και οι προδιαγραφές ζωής σημαίνουν ε, και η υγιεινή διατροφή. Στην Ρουμανία έχουμε πολλούς γεωργούς, αλλά τα αγροκτήματα είναι πολύ μικρά. Τι στήριξη θα δώσετε στους μικρούς γεωργούς, ιδιαίτερα στα νέα κράτη-μέλη. Σας ευχαριστούμε. Υπουργέ, με στα νέα κράτη-μέλη έχουμε διαφορετικού όρους και προποθέσει, Για παράδειγμα, στη χώρα μου που δεν έχει τόσε πολλές μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσει όσο, όσο υπάρχουν αλλού σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Έχουμε μια πολύ ανταγωνιστική γεωργική βιομηχανία και σε μεγαλύτερη κλίμακα. Όταν όμω πάει κανεί στην κοντινή Πολωνία η κατάσταση είναι διαφορετική εκεί. Τώρα το ζήτημα το οποίο θέτει η κυρία Ντόιλ με την ερώτησή της ε, τι κάνουμε ακριβώς. Έχω κάποιους γεωργούς ε, στην ε, δική μου εκλογική περιφέρεια στη Βοημία. Τα πάνε καλύτερα επειδή έχουν περισσότερα κονδύλια. Έχουμε και γεωργούς που έχουν χειροστάσια δεν υπήρχε αυτή η διαμόρφωση αυτής της κατάστασης πριν από μερικά χρόνια. Ταυτόχρονα όμως αισθάνονται ότι υφίστανται κάποια αδικία λόγω του διαφορετικού επίπεδου πληρωμών μεταξύ των παλαιότερων κρατών μελών και των νεότερων κρατών μελών. Είναι θέμα θεμελιώδους δικαιοσύνης που θα έπρεπε να εισαχθεί στο σύστημα. Πρέπει να επαναρθωθεί λοιπόν το διαφορετικό επίπεδο πληρωμών. Και ταυτόχρονα πιστεύουμε ότι η ΚΑΠ θα έπρεπε να μεταρρυθμιστεί. Είναι ο μόνος λοιπόν τρόπος για να επιτευχθεί ο στόχος της ανταγωνιστικότητας, της βελτίωσης της Ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητας στην Γεωργία. Έχουμε εδώ ένα σύνθετο πρόβλημα, δεν επισέρχομαι σε λεπτομέρειες, όμως τουλάχιστον οι βασικές ε, κατευθυντήριες γραμμές είναι σαφείς και πρέπει να συμφωνήσουμε από αυτόν. Ευχαριστώ. Κυρία Τικάου για το ερώτημά. I'm ευχαριστώ. Λυπάμαι συνάδελφοι, αλλά σήμερα προβλέπετε να κλείσουμε στις 8. Οπότε οι ερωτήσεις 6 μέχρι και 29 θα απαντηθούν γραπτός. Και έτσι τελειώνουμε τις εργασίες μας. Ευχαριστώ τον Υπουργό και κλείνει η συνεδρίαση μέχρι τις 9 το βράδυ.